ο προηγούμενος ε, επίτροπος ε, της ΑΝΚΟ μας είχε διαβεβαιώσει ότι όχι μόνο θα εφάρμοζε την παρούσα νομοθεσία σωστά, αλλά ότι θα, θα αναθεωρούσε την ε, κατάσταση, θα έκανε έναν έλεγχο επαναμία με επανεξέταση της όλης κατάστασης μέχρι το τέλος της θητείας μας. Τελειώνει όμως αυτή η κοινοβουλευτική θητεία, τελειώνει και η θητεία της Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να απευθύνω μια έκκληση στην κυρία Βασιλείου, η οποία ήταν ανάξια διάδοχο του κύριου Κυπριανού, να υιοθετήσει τις δεσμεύσεις του κυρίου και να σεβαστεί τις δεσμεύσεις του κυρίου Κυπριανού, διότι η μεταφορά των ζώων είναι από τα θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν αυτά, αλλά είμαστε μια πολιτισμένη κοινωνία και μια πολιτισμένη κοινωνία πολλές φορές κρίνεται όχι μόνο από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους ανθρώπους αλλά και με τον τρόπο με ε, τον, με τον οποίο ε, χειρίζεται τα ζώα. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Τώρα, για την προφορική ερώτηση αυτή καθεαυτή. Η μεταφορά, ο κανονισμός για τη μεταφορά των ζώων ε, είναι σε ισχύ από το 2005 η Κομισιόν έπρεπε να, πάει, να έχει πάρει τουλάχιστον την πρώτη ετήσια έκθεση από τα κράτη-μέλη σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Μπορεί η Κομισιόν να μας πει ποια είναι τα κράτη-μέλη έχουν υποβάλει την έκθεσή τους η Κομισιόν έχει κάνει ήδη μια προκατακτική ε, ανάλυση ενδεχόμενα, επομένως θα έχει μια γενική εικόνα για τα μειονεκτήματα, για για τα προβλήματα, για τα κενά Επομένως, μήπως θα μπορούσε η Κομισιό να μας πει ποια, πώς έχει, ποια είναι, πού βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς του κανονισμού στα κράτη-μέλη. γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε κάπως τον κανονισμό για τη μεταφορά των ζώων με βάση τα διδάγματα από, τις, από την εμπειρία μας μέχρι τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Κομισιό, ο κύριος Σπίτλα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ απολύτως με την άποψη του κυρίου Πάρης ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα ζώα συμπεριλαμβανομένων και των ζώων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, είναι θέμα ηθικής και διοντολογίας καθώς και ένδειξη πολιτισμού. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι η μεταφορά ζώων για εμπορικούς σκοπούς ε, μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία και μάλιστα σημαντική ταλαιπωρία στα ζώα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζώα που θεωρούνται χαμηλής αξίας, δηλαδή τα ζώα που προορίζονται για σφαγή. Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα τα οποία ισχύουν ε, για την ε, μεταφορά ζώων ε, και μάλιστα σε μακρές αποστάσεις και έχουμε ακούσει αναφορές για κακή μεταχείριση των ζώων και θέλουμε να εφαρμόσουμε το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσουμε και την υγεία των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Σε μια μελέτη που έγινε από το, κέντρο, από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται καλύτεροι τρόποι ελέγχου, όπως ε, παρακολούθηση και μέσω δορυφορικού συστήματος, για να εντοπίζονται γεωγραφικά οι διαδρομές ε, μεταφοράς των ζώων θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση. Θέλουμε επίσης να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και για τις εθνικές και άλλες αρχές. Αξιολογεί ακόμη η Επιτροπή την ε, δυνατότητα μέχρι το τέλος της θητείας μας ε, να προτείνουμε νέους κανόνες και προδιαγραφές βάσει της ισχύουσας επιστημονικής γνώσης για το για τη χρονική διάρκεια των μεταφορών και για τον αριθμό των ζώων αναόχημα. Η Επιτροπή βασίζεται στις εκθέσεις των κρατών μελών για την αξιολόγησή της, εκθέσεις που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού που ισχύει αυτή τη στιγμή. και οι εκθέσεις αυτέ βασίζονται σε κτηνιατρικού ελέγχους που έχουν γίνει στα κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών δημοσιεύεται στις ιστοσελίδε της Επιτροπής και γίνεται η αξιολόγηση συγκρίνοντας τις πληροφορίες και με πληροφορίες μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη υποβάλει τις εκθέσεις τους για το 2007. Μέχρι το τέλος του 2008 η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν υποβάλει ακόμη έκθεση. Πράγμα το οποίο έχει επισημάνει η Επιτροπή και θα παρακολουθούμε την κατάσταση επαγρυπνώντας. Ο κανονισμός 1 του 2005 πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη και η επιβολή της νομοθεσίας είναι βασικό στοιχείο κάθε νομοθεσίας και τώρα και στο μέλλον. Και γι' αυτό η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις αναλύσεις των κρατών μελών με στόχο την περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Στίβενσον θα πάρει το λόγο εξ ε, του Λαϊκού Κόμματο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρα και Επίτροπε κύριε Σπίδλα. Θα ήθελα, ας δούμε λίγο ε, ποιο είναι το υπόβεθρο της όλης της ιστορίας. Είχαμε 8 ώρες για την μέγιστη μεταφορά των δι... Ε, των, κρατών, των ζώων ή τη μεταφορά των ζώων. Αυτό και σε, ε, υιοθετήθηκε το 2005 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2007. Βέβαια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εφαρμόστηκε αυτό, διότι έπρεπε να προσαρμοστούν οι τεχνικέ προδιαγραφέ των ζώων, αν υπήρχε κλιματισμός, αν υπήρχε εξαερισμός ε, και γενικότερα ε, ε, δόθησαν και κάποιε εξαιρεσει για κάποιε απομακρυσμένε περιοχέ τη υπαίθρου ή νησιά. Σε, εμά α πούμε, στη χώρα μου, στο Κλί και στα Σέτλαντα όμως υπήρχε, έπρεπε να σχεδιαστούν και οι κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο νερό και τα ζώα να ταξιδεύουν με κάποια άνεση. Για κάποια ε, ζώα όμως υπήρξε απόλυτη απαγόρευση για, τις, για τα μοσχαράκια ε, μέχρι 10 ημερών και αρνάκια μέχρι μιας βομάδας. Μπορώ να σας πω ότι ε, σε περιοχές όπως η Σκοτία οι μεταφορές παρακολουθούνται πάρα πολύ προσεκτικά και ε, στη Σκοτία έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα καλύτερων πρακτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όπως και μας είπε και ο Νίλ Πάρις, με ανησυχούν κάποιες ε, πληροφορίες που λένε ότι δεν γίνεται η σωστή παρακολούθηση σε άλλα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη στι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα νέα κράτη. Και όπως είπε και ο Νίλη Πάρη, όταν, κυρίως όσον αφορά την μεταφορά των αλόγων για σφαγή οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, διάφορες ε, άλλες ε, οργανώσεις παρουσιάζουν στοιχεία για τις μεταφορές των αλόγων κάτω από τραγικές συνθήκες, μεγάλες διαδρομές χωρίς νερό, χωρίς εξαρισμό, χωρίς ανάπαυση και όσο προχωράει το ταξίδι εξαντλούνται και αφιδατώνονται τα άλογα, τα ζώα αυτά, υποκύπτουν ε, στο στρες της ζέστης, ε, δεν μπορούν να αναπνεύσουν και πολλά ζώα πεθαίνουν στο τέλος. Αυτά είναι πράγματα, αυτή είναι μια πρακτική η οποία πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να γίνεται σεβαστά, σεβαστή απόλυτα η νομοθεσία. Επομένως, ε, συμφωνώ απόλυτα με την προφορική ερώτηση του Νίλ Πάρις, διότι θα πρέπει να ελέγξουμε το επίπεδο συμμόρφωσης με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί και νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να μας δώσει τις ε, κατάλληλες πληροφορίες και να μας πει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε οι 8 ώρες μέγιστη διάρκεια ταξιδιού να γίνουν σεβαστές. Και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την σκληρή παραβίαση ε, της κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, η κυρία Μιγγέλες Ράμους. Κυρίες και κύριοι, για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είπε ο κύριος Στίβενσον, για γεωγραφικούς λόγους ή λόγω του μεγέθους της επιφανίας τους ή για λόγους εμπορίου, παίζει ιδιαίτερο ρόλο η μεταφορά των ζώων. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημαντικά σημεία, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι είναι προφανές ότι η Επιτροπή ακόμη έχει προβλήματα στην καταγραφή της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι σύμφωνα με τον τωρινό κανονισμό τα κράτη-μέλη πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλουν έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι έρευνες που έγιναν κατά το παρελθόν έτος, ο κανονισμός δεν ορίζει ελάχιστο αριθμό ερευνών που πρέπει να έχουν γίνει, ούτε μιλά για κάποια στατιστική βάση. Άρα τα δεδομένα τα οποία δίδουν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συγκριθούν ε, μετά τη συλλογή τους. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Με ανησυχεί επίσης και άλλο ένα σημείο. Στην ομιλία σας, ε, κύριε Επίτροπε, Αναφερθήκατε στα ζώα τα οποία πηγαίνουν προς σφαγή και είπατε ότι είναι χαμηλής οικονομικής αξίας. Εγώ διαφωνώ. Είναι υψηλής οικονομικής αξίας και νομίζω ότι και ο σχετικός τομέας, ο σχετικός κλάδος θα συμφωνήσει μαζί μου. Είναι μεγάλη οικονομική τους αξία και για να διασφαλίσουμε την υψηλή του αξία θα πρέπει να τους διασφαλίσουμε σωστές συνθήκες μεταφοράς, όποια και αν είναι η απόσταση στην οποία θα μεταφέρονται. Θα πρέπει λοιπόν τα ζώα αυτά να μεταφέρονται σε σωστές συνθήκες και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές στον κανονισμό. Αυτή η μεταρρύθμιση του κανονισμού ξέρουμε ότι θα συμπεριλαμβάνει κάποιες ε, τροποποιήσεις σχετικά με το μέγιστο χρόνο μεταφοράς, σχετικά με τον ελάχιστο και μέγιστο ε, βαθμό θερμοκρασίας και ζητώ από εσά κύριε Επίτροπε, ζητώ από την Επιτροπή, πριν κάνετε τέτοιες μεγάλες τροποποιήσεις, να φροντίσετε να έχετε την κατάλληλη επιστημονική βάση για να μπορέσετε να βασίσετε τη σωστή μεταρρύθμιση. Σε πολλά σημεία δεν έχουμε ακόμη ε, επιστημονικά δεδομένα. Τα επιστημονικά δεδομένα θα χρησιμεύσουν ως βάση ούτως ώστε να μην παρισφύγουν ε, κάποιες διατάξεις που θα επιτρέπουν ε, εσφαλμένη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους. Θα πρέπει να παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Τζένσεν εξ ονόματος των, των, Μπορώ να σας πω ότι μετά από τέσσερα χρόνια είμαι κάπως απογοητευμένη διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευρά τη Κομισιόν για να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία υπάρχουν καλές προθέσεις, υπάρχει μια ε, καλή συνεργασία ανάμεσα στην κυρία Βασιλείου και στο Κοινοβούλιο. Αποτέλεσμα όμως μηδέν. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και χρειάζεται μία εγγύηση ότι θα περιοριστεί σε 8 ώρες η διάρκεια της μεταφοράς των ζώων. Δεν θα πρέπει όμως να μιλάμε μόνο για τη διάρκεια, διότι οι αποδείξεις είναι μπροστά μας ότι ακόμα και μία ώρα ταξιδιού μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα αποδυναμωμένο ζώο ενώ ένα ζώο σε καλή υγεία και κάτω από καλές συνθήκες μπορεί να μεταφερθεί ίσως και παραπάνω από 8 ώρες. Όμως εδώ μιλάμε για ε, μεταφορές που είναι ε, σε, ε, σε μεγάλες αποστάσεις και χρειάζονται, χρειάζονται πάνω από 24 ώρες για τη μεταφορά τους. Επομένως, τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει οι κτηνίατροι, οι διάφορες οργανώσεις, ε, οι μεταφορείς να ε, συγκεντρωθούν κάπου και να αποφασίσουν για τις καλές πρακτικές. Αυτές, αυτές οι πρακτικές πρέπει να εφαρμοστούν και θα πρέπει να μεταφερθούν και στην νομοθεσία. Ο κύριος Βοητσεκόφσκι για ένα λεπτό. Πολύ σωστά. Το είναι μια σκέψη την οποία να έχουμε ε, σκεφτεί και εμείς ε, εδώ ε, και το έχουμε ξαναπεί και στην Ολομέλεια ότι οι συνθήκες, αυτής μεταφο... αυτές μεταφοράς δείχνουν το πολιτισμικό μας επίπεδο. Θα πρέπει ε, να ανέβουν, έχουν ανέβει αρκετά τα στάνταρτς και οι προδιαγραφές, όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και οι προδιαγραφές αυτές. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να περιοριστεί η μέγιστη διάρκεια ε, της μεταφοράς σε 8 ώρες. Επίσης, η, ο χρόνος στον οποίο περνάνε τα ζώα στο σφαγείο θα πρέπει να περιοριστεί ε, στις 12 ώρες κατά μέγιστον. Ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο προσπαθούμε, το προσπαθούμε όλοι μας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει γενικώ να περιορίσουμε τις μεγάλες μεταφορές, διότι οι μεγάλες αυτές μεταφορές των ζώων ε, αυξάνουν το κόστος του κρέατος και επομένως θα πρέπει να περιορίσουμε και την μεταφορά για να περιορίσουμε και την αγωνία των ζώων. Ο κύριος Σλίτερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισμού μπορεί να μετρηθεί με τον τρόπο κατά τον οποίο μεταχειριζόμαστε τους πλέον αδυνάτους και εμάς θα μπορούσε να μας χαρακτηρίσει κανείς βαρβάρους αν κρίνει από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα ζώα. Η Σουηδία είναι τώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την ένταξή της ε, είχε διαπραγματευτεί τα θέματα βελτίωσης ε, της ε, μεταχείρισης των ζώων. Υπήρχε ο κανονισμός του 2005. Στη συνέχεια είπαμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, ενδεχομένως και με ένα σύστημα GPS για να έχουμε πληροφορίες για την ε, μεταφορά των ζώων. Και πέντε, χρο... πέντε χώρες δεν έχουν καν υποβάλει την έκθεσή τους. Χρειάζεται λοιπόν η Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα. Πώς λειτουργεί αυτή η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Λειτουργεί ο κανονισμός σωστά. Δυστυχώς η απάντηση είναι όχι. Ο κύριος Κυπριανού μας είχε υποσχεθεί κάτι. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί μέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής. Και μπορεί ο χρόνος μεταφοράς να μειωθεί γιατί είναι πολλές οι χώρε που είναι μικρές και επομένω δεν χρειάζονται μεγάλο χρόνο μεταφοράς ε, των ζώων. Υπάρχουν και κινητά σφαγεία οπότε μπορεί να συντομευθεί ο χρόνος ε, ε, μεταφοράς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή και για, για πολλά ζώα, για τις αγελάδες, για τα κοτόπουλα. Κανείς δεν θα ήθελε να υφίσταται τέτοια μεταχείριση. Όλοι οι υπουργοί μεταφορών θα έπρεπε να μεταφερθούν από τη Σουηδία μέχρι το κέντρο της Ευρώπης στις ίδιες συνθήκες με τα ζώα για να καταλάβουν πόσο τραγικές είναι οι συνθήκες. Το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό διότι η απόσταση μεταφοράς είναι μεγάλη, αλλά μας ενδιαφέρει η σωστή ποιότητα της μεταφοράς για να είναι καλύτερες οι συνθήκες ε, διαβίωσης των ζώων και καλύτερη η ποιότητα του κρέατος, γιατί αν ένα ζώο ταλαιπωρείται, λόγω της πίεσης την οποία υφίσταται και το κρέας του είναι χειρότερης ποιότητας. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια απάντηση της Επιτροπής που θα εγγυάται την βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς των ζώων για να κάνουμε και εμείς μια προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Χόλμ για τρία λεπτά. Για δύο λεπτά, συγγνώμη. Εξ ονόματος της Γκουε. Κοιτάξτε, τα ζώα αισθάνονται τον πόνο και το στρες υποφέρουν ακριβώς όπως και οι, άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν ε, ε νομοθετούμε. Αυτό δεν το έχουμε κάνει τώρα. Εδώ όλο ένα και περισσότερα ζώα μεταφέρονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια συνέπεια της εσωτερικής αγοράς. Αλλά και έχει γίνει μια φοβερή εξειδίκευση. Τα ζώα εκτρέφονται σε ένα σημείο, μεταφέρονται σε ένα άλλο όπου εκεί σφάζονται και μετά υπάρχει και μεταφορά σε ένα τρίτο σημείο που γίνεται η επεξεργασία τους και η μεταποίησή τους. Θα πρέπει να κάπως να τα, να τα ομαδοποιήσουμε αυτά. Μία μελέτη που έγινε στη Σουηδία με, προσπάθησε να μετρήσει την ε, μεταφορά της διελεύσης των ζώων ε, από τα σύνορα. 22 εκατομμύρια ζώα περνάνε τα σύνορα. Και 500 εκατομμύρια ε, κοτόπουλα. Αυτός είναι ο αριθμός για την Ευρώπη των 15. Και ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, η νέα οδηγία για την, μετα... τη νέα οδηγία για την μεταφορά των ζώων, πότε θα την έχουμε. Ο κύριος Κυπριανού μας την είχε υποσχεθεί για αυτή τη θητεία. Υπάρχει περιθώριο να περιμένουμε τώρα, να έχουμε δηλαδή αυτό το όριο των 8 ωρών. Και ο κύριος Σπίτλα μίλησε για τα για αυτά τα πέντε κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υποβάλει την ετήσια έκθεσή τους. Αυτό είναι σοβαρό. Αλλά από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν υποβάλει τις ετήσιες εκθέσεις τους. Αυτές τις εκθέσεις τις έχετε αναλύσει. Εμείς χρειαζόμαστε, πιστεύω, μια συγκριτική ανάλυση όλων αυτών των εκθέσεων για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με τη μεταφορά των ζώων. Λοιπόν, δύο πράγματα νέα οδηγία και η ανάλυση των ετησίων εκθέσεων που έχουν βάλει τα κράτη-μέρη. Ο κύριος Μπλουμ για δύο λεπτά. Well, Κύριε Πρόεδρε, είναι πάντοτε συνεργαστικές συζητήσεις που γίνονται στην Ολομέλεια. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ανοησία των κανονισμών που δόθηκαν στα σφαγεία πριν από 10 χρόνια που είχαν ως αποτέλεσμα το να κλείσουν πάνω από χίλια σφαγεία και τελικά παρέτειναν την ε, ε, διάρκεια μεταφοράς των ζώων. Ο γαμπρός μου είναι ε, χασάπης και μου λέει ότι κάποια φορά υπήρχε κάποιος ο οποίος επέβλεπε ένα κτηνίατρο, ο οποίος επέβλεπε κάποιους υπαλλήλου που επέβλεπαν τη διαδικασία σφαγή. Νομίζω ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τέτοια γραφειοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγαλύτερου χρόνου μεταφορά, γιατί από τη δική μου εκλογική περιφέρεια πρέπει να φτάσουν στο Μάντσεστερ τα ζώα για τη σφαγή τους λόγω ακριβώς ε, του κανονισμού που επέβαλε το κλείσιμο των σφαγείων που σας ανέφερα. Επίσης μας ανησυχεί και το θέμα της μεταφοράς ε, των αλόγων. Ο συνάδελφος Νάιτζορ Φεράς μου λέει ότι σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα άλογα θεωρούνται φαγητό. Εμένα μου φαίνεται τραγικό αυτό. Για μας τους Άγγλους είναι τραγικό το να τρώει κανείς το άλογό του. Δεν θα τρώγαμε το άλογό μας όπως θα τρώμε το γιο μας και την κόρη μας. Αυτό δείχνει την τεράστια πολιτιστική διαφορά, το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ημών και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους μη εγκεκραμένους, ο κύριος Άλιστερ για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το να ακολουθήσω μετά από όσα ακούστηκαν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία δυσκολία να έχουμε αποτελεσματικούς και σωστούς κανόνες που να διέπουν την ευημερία των ζώων. Όμως ανησυχώ γιατί νομίζω ότι μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο. Θα ε, κάνουμε τόσο αυστηρούς τους κανόνες και θα δέσουμε τα χέρια της των γεωργών που δεν θα είναι δυνατόν να αποδώσουν. Και βλέπω τέτοιου είδους ε, δείγματα ε, από τις διαβουλεύσεις με την, Κομισιό, με την όσον αφορά την αναθεώρηση της μέγιστης διάρκειας και την ε, αναθεώρηση της πυκνότητας των ζώων μέσα στα φορτικά. Η Κομισιό υιοθέτησε βοήθησε να υιοθετηθεί ο κανονισμός το 2005. Όμως τρία χρόνια μετά προσπαθούν αφαιρώντας την προσπαθούν ακόμα περισσότερο υιοθετώντα αυτό το μέτρο των, ή θέλουν να υιοθετήσουν το μέτρο των 8 ωρών. Για μας θα είναι καταστροφικό, διότι για να εξάγουμε τα ζώα απαιτείται μεταφορά διαθαλάσσης. Και αν έχουμε 8 ώρες, αυτό δεν θα, δεν θα αρκέσει. Θα δηλαδή είναι δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και τόσο βεβαρημένες συνθήκες, πρέπει να σας υπενθυμίσω, ότι δεν συγκρίνονται κατ' ουδέναν τρόπο με τις τεράστιες αποστάσεις που πρέπει να μεταφέρονται τα ζώα στην Νότια Αμερική, από την οποία χωρίς κανένα πρόβλημα εισάγουμε κρέατα. Επομένως, για άλλη μια φορά τιμωρούμε τους δικούς μας αγρότες χωρίς να, σεβα... χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις συνέπειες των εισαγωγών. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι θα πρέπει <clears throat> κάποια στιγμή να μην ε, ε, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα να κάνουμε ε, μόνοι μας, να με βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση και να καθησυχάσω τον κύριο Μπλουμ όσον αφορά την ε, κατανάλωση του ε, κρέατος των αλόγων ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να σας πω να σας πω ότι ναι μεν καταναλώνεται κρέας αλόγου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κανείς καταναλωτής δεν θα φάει το δικό του άλογο. Θα φάει το άλογο ενός άλλου. Λοιπόν, η κυρία Γέγκλε για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητάμε ένα θέμα στο οποίο βλέπει κανείς ε, ότι πολύ γρήγορα ε, υπάρχουν πολλά συναισθηματικά στοιχεία και υπάρχουν, ε, υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα από την άλλη πλευρά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω για συναισθήματα. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα, κύριε Επίτροπε, τι έχει γίνει. Έχετε εκθέσεις, έχετε στοιχεία, τι αριθμητικά στοιχεία έχετε. Έχετε στοιχεία που θα μας οδηγούσαν σε ένα αποτέλεσμα που θα δείχνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ κρατών μελών. Μια βασική διαφορά είναι ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν υποβάλει έκθεση, κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν υποβάλει έκθεση. Πώ γίνεται ο έλεγχο των μεταφορών σε κάθε κράτο μέλο, σε ποια κράτη-μέλη υπάρχει ηλεκτρονικό έλεγχο. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε επιγόντως ε, είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στον τομέα της γεωργίας και που έχουν σχέση και με τον οικονομικό τομέα ε, και εδώ υπάρχει πολύ συχνά διαφορετική αντιμετώπιση. Για τις ε, μεταφορές των ζώων τι κατάρτιση πρέπει να έχει ο υπεύθυνο ε, της γεωργικής εκμετάλλευσης, τι αποδεικτικά κατάρτισης χρειάζονται. Πώς έχει εκπαιδευτεί αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ε, μεταχείριση των ζώων. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καν υποχρέωση ε, κατάρτισης. Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Και άλλο ένα πρόβλημα είναι όταν ε, ένας ε, αγρότης μεταφέρει ε, τα δικά του ζώα, μπορεί να τα μεταφέρει μέχρι απόσταση 50 χιλιόμετρων. Αυτό θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν κάποια μικρά σφαγεία στην γειτονική περιοχή για να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες αποστάσεις. Αν όμω ο γεωργό εκτό από τα δικά του ζώα θέλει να μεταφέρει και τα ζώα του γείτονά του, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό τα 50 χιλιόμετρα είναι πραγματικό όριο. Πρέπει να δούμε πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στα κράτη-μέλη για να δούμε τι τροποποιήσει χρειάζονται. Υπάρχουν επίση ε, και οι περιπτώσει μεταφορά ζώων, μεταφορά αλόγων ε, για λόγους αναψυχής και όχι για ε, λόγους γεωργίας. Είναι και αυτό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της Επιτροπής και πρέπει να έχουμε τα στοιχεία αυτά για να μπορούμε να κάνουμε τη σωστή συζήτηση. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά έχει τώρα το λόγο ο κύριος Καπούλας Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε τώρα το θέμα τη μεταφορά και τη χρονοταχείριση των ζώων, που είναι ένα ζήτημα το οποίο πάρα πολύ σωστά ε, είπαν οι προελίσσαντε. Θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και από πλευρά πολιτισμού. Είναι μια επιταγή ηθική το να φερόμαστε καλά στα ζώα. Είναι κάτι το οποίο χειρίζεται στον πολιτισμό, στην κουλτούρα μας. Άλλωστε, λέμε τώρα για την κατανοχήρησή του στο τελευταίο του ταξίδι. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτές οι διατάξεις, αν ε, εφαρμοστούν, ε, θα κοστίσουν. Και λέγεται βέβαια ότι για κάποιες περιφέρειες, για βιάκαρα κάτι μέλη, ε, θα βαρύνει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό αφορά και τη δική μου χώρα θα έχουμε δυσκολίες να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό θα αφορά και τη μεταποίηση. Θα αποκτήσουμε επομένως μειονέκτημα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ε, έχουν καλύτερη δυνατότητα το να μεταφέρουν τα προϊόντα, ε, να τα περάσουν από τη μεταποίηση και κατόπιν να τα πουλήσουν σε πιο ανταγωνιστική τιμή. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει και να ζυγίσει όσο γίνεται καλύτερα ε, όχι μόνο τα στενά θέματα εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία, αλλά να κάτσουν και να μελετήσουν ποιε θα είναι οι κοινωνικέ αλλά και οι οικονομικέ συνέπειε για τι διάφορε περιφέρειε, για διάφορα κράτη-μέλη, ε, εκεί όπου ε, υπάρχει πρόβλημα, είναι η η παραγωγή κάποιων ε, ζώων που είναι πάρα πολύ βασικά για την εκτινοτροφία. Όλα αυτά πρέπει να τα δείτε όσο πιο βαθιά γίνεται. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Ντίρτσαρ Μούρκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Η Σλοβενία είναι χώρα από την οποία παίρνουν πάρα πολλές μεταφορές ζώων και από την ε, Ιταλία κυρίως ε, έχουμε τέτοιες μεταφορές που διασχίζουν τη χώρα μας. Επομένως θα πρέπει να δούμε πως ε, όλο αυτό το πλαίσιο των διατάξεων που υπάρχει θα είναι πιο ευέλικτο ούτως ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα. Να δούμε τι θα γίνει και με τις επιθεωρήσεις τους ελέγχους. Γιατί έχουμε μεν κατάρριξη των εσωτερικών συνόρων, όμως είναι δύσκολο να ελέγξουμε αν και πού σταμάτησαν ε, τα φορτηγά. Πού έκαναν στάση οι οδηγοί. Βέβαια και λόγω της, ε, του, του μεγέθους της χώρας μας ε, έχουμε σχετικές συμφωνίες με Ουγγαρία και Ιταλία. Άρα θα πρέπει να μια αποδοτική, μια, μια λύση που να αποδώσει αποτελέσματα και έτσι να υπάρχει περισσότερη καλομεταχείριση στα ζώα όταν διασχίζουν τους ευρωπαϊκούς δρόμους και αυτή η νομοθεσία του 2005 θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μεταφορά των ζώων φυσικά ε, και έχει να κάνει με το πώς μεταχειριζόμαστε τα ζώα πριν πάνε στο σφαγείο. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι δεν θα πρέπει να έχουμε διαδρομές μεγαλύτερες των 8 ώρων. Εγώ σας προτείνω να υπάρχει ένα τέτοιο ανώτατο όριο και επίσης να δούμε τι θα γίνει με τα κινητά σφαγεία. Σαπαλόφσκι. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε αυτόν τον κανονισμό που αφορά τη μεταφορά των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα και επίσης ε, κάθε φορά η άντληση των σχετικών πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Άλλωστε τελικά οι Ευρωπαίοι πολίτες καταναλώνουν αυτά τα ζώα. Όμως ε, λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για αξιόλογο νομοθέτημα το οποίο αφορά την ευημερία των ζώων και αλλά και το νομοθέτημα που αφορά τις συνθήκες σφαγής. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, πάρα πολύ προσεκτικά αυτή η νομοθεσία και άλλωστε μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχουν πρόβλημα εφαρμογή των νομοθεσιών για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα με τα ζώα. Οι ιδιωτικές αρχές επίσης θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι διατάξεις. Σύνοτ, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, πάρα πολύ σημαντικό είναι το, το να έχουμε ασφαλή μεταφορά των ζώων, να μην υπάρχει αχρίαστη ταλαιπωρία των ζώων και έτσι κι αλλιώς δεν αρέσει τα ζώα αυτή η μεταφορά, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία τους, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, συνήθως έχουμε ως κριτήρια την απόσταση αλλά και τον χρόνο μεταφοράς. Αυτό είναι λογικό, αλλά από την άλλη μεριά είναι απλουστευτικό, γιατί όσον αφορά την περίπτωση της Ιρλανδίας, το πρώτο έχουν άλλο, μια που είμαστε ένα νησί και άλλωστε είμαστε και μέγας εξαγωγός κρέατος, οπότε έτσι κι αλλιώς θα πρέπει εμείς να διασχίσουμε τη θάλασσα της Ιρλανδίας για να φτάσουμε στην αγορά. Ε, αυτές οι 8 ώρες που τάσσονται ως όριο δεν, δεν, δεν κολλάνε στη μας περίπτωση ε, τόσο να διασχίσουμε τη θάλασσα για να φτάσουμε στην ε, αγορά. Ούτε είναι δυνατόν φυσικά κανένα να σταματήσει μέσω πελάγου και να βάλει τα ζώα να κάνουν μια βόλτα και να βοσκήσουν άλλα. Άρα θα πρέπει περισσότερο να δει κανεί υπό ποιε συνθήκε γίνεται η μεταφορά πέραν του, του, του στενού κριτηρίου, τη απόσταση αλλά και του χρόνου. Ο πρόεδρο. Και δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός για την μεταφορά των ζώων έχει τεθεί σε ισχύ από τον Γενάρη του 2007. Φαίνεται όμως ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί υποβάλλοντας τις ετήσιες εκθέσεις που, προ... που προβλεπόντουσαν. Επομένως, μία ανάλυση ενδελεχής δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά τις, ε, τους... και πρέπει να γίνουν διάφοροι έλεγχοι κτλ. Ε, διάφορες ε, διοκομματικές οργανώσεις έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Οι ενώσει δίνουν μία άνεση μάχη εδώ και 10 χρόνια για να καταφέρουν ε, τουλάχιστον το 2007 να υιοθετηθούν κάποιε οδηγίε ε, για τα θέματα αυτά, διότι υπάρχει μια χαλαρότητα από πλευρά των κρατών μελών, για να μην πω και μια κακή θέληση. Γιατί το ξέρουμε ούτως ή άλλω ότι η αλλω οτι η εφαρμογη των ελέγχων και και των επιθεωρήσεων δεν είναι ένα εμπόδιο ανυπέρβλητο. Ξέρουμε πού, πού είναι τα σφαγεία, πού ε, εκτρέφονται τα ζώα, ε, πού είναι το πρόβλημα τότε. Ε, αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, όπου η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και πολύ σωστά για την κατάσταση των ζώων, είτε πρόκειται για την κατάσταση των σφαγείων, είτε κατάσταση των, της μεταφοράς, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις διατάξεις τις νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, μια και έχω το λόγο να σας πω ότι είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε και να λάβουμε υπόψη μας ανεξάρτητα από τη διάρκεια των μεταφο... της μεταφοράς και τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, μία μεταφορά που διαρκέστο και πολλές ώρες ε, την άνοιξη το στις κάτω χώρες δεν έχει καμία σχέση με την, και δεν, δεν, δεν υπάρχουν, ε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια πράγματα όπως με μια μεταφορά το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ο πλευράς της νομοθεσίας τώρα μιλούμε για έναν σχετικά νέο κανονισμό τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2007. Όλοι ελπίσαμε ότι αυτές εξ αρχής θα συμμορφωθούν όλοι μετά όσο επιτάσσει ο Όμως αυτό μάλλον ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρός αυτός ο οικονομισμός και για τα κράτη και για τους ε, εμπορευόμενους. Πάρα πολύ σωστά το είπε ο κύριο Πάρη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να αποδώσει αυτό ο αγωνισμό, να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί. Γιατί μα ενδιαφέρει το πώ μεταφέρονται τα ζώα. Ε, Εμεί, όπω ξέρετε, έχουμε εκτεταμένη κτηνοτροφία στην Ιρλανδία και έχουμε πάρα πολύ σκληρά δουλέψει τόσο ώστε να εφαρμοστεί ο κανονισμό και οι αρχέ και οι κτηνοτρόφοι. Και έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικέ ε, επενδύσει τόσο ώστε η μεταφορά να γίνεται όπως πρέπει, να εκπαιδευτούν οι οδηγοί κλπ. Ήδη αυτό το μήνα για τους οδηγούς των φορτηγών που μεταφέρουν τα ζώα, όλα τα ζώα, γίνεται ένα σεμινάριο εκπαιδευτικό. Ε, όπως είπε η κυρία Γέγκλε, θα πρέπει να μας μιμηθούν και οι άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει βέβαια να εξεταστεί και το τι συνέπειε θα έχουν όλα αυτά για την οικονομική δραστηριότητα. Θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται με τα κατοικίδια ζώα. Και εκεί δεν νομίζω ότι ε, ο κόσμος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Προσοχή γιατί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που κακομοιρίζουν τα δικά τους ζώα ε, γκρινιάζουν για την κτηνοτροφία υπάρχει ένα πλαίσιο έγκρισης ε, και αδειοδότησης για τη μεταφορά των ζώων και έλεγχος ούτως ώστε τα ζώα να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή όπως πρέπει. Θα πρέπει επομένω ε, όλοι στον κλάδο να εφαρμόσουν τον ε, κανονισμό, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του και όποιος το κάνει οι κυρώσεις να είναι πάρα πολύ αυστηρές, να τον πετάμε έξω από το κύκλωμα. Βέβαια, ε, εμεί λόγω γεωγραφική θέση ε, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μεταφορά των ζώων, αλλά ξέρουμε και τι να κάνουμε. Ε, οπότε, εντάξει, να μην συρρυκνωθούν τα όρια τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά να είναι πιο ευέλικτε διατάξει όσον αφορά την ποιότητα τη μεταφορά. Επίσης κάποιες φυλές ζώων αξίζουν περισσότερο από άλλες. Ε, αυτό αφορά και τα καθαρό άλογα και εκεί θα πρέπει να έχουμε κάποιες ε, σωστές διατάξεις. Όμως προσοχή η πολυνομία να μην φέρει ασφυξία στον κλάδο. Όμως ό,τι διατάξεις και να υπάρχουν να ισχύουν για όλους και όποιος τους εφαρμόζει να τον πετάμε έξω από το σύστημα Evans. Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Πάρης για τις προτάσεις του, παρά το ότι έχουν πολιτικές διαφορές. Ε, νομίζω ότι παρά όλα του τα κουσούρια, τα ανθρώπινα, πάρα πολύ σωστά τα είπε εν προκειμένου. Χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό, χρειαζόμαστε να εφαρμοστεί επιτυχώς και να εφαρμοστεί παντού. Εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και διαφωνώ με κάποιους από αγορεύσαν τους συναδέλφους. Ο κύριος Στίβενς είπε ότι είναι αναπόφευκτα κάποια ταξίδια μεγάλα, διαφωνώ, είπατε για 24 ώρες κυρία Γιάγκλε, ούτε αυτό είναι αναγκαίο, αναγκαστικό να συμβαίνει. Για τον κύριο Μακάλιστερ επίσης και εκεί διαφωνώ στα όσα είπε, θα πρέπει επομένω όλοι ως κοινωνία να δούμε αυτό το θέμα καλύτερα τις μακρές αυτές μεταφορές και κατόπιν τη σφαγή των ζώων. Να μην υποφέρουν τα ζώα, να μην υφίστανται αφιδάτωση, αγωνία. Ε, όλοι, όλοι να σε βορρά και σε νότο θα πρέπει να εξετάσουμε πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση ούτως ώστε και το τελικό προϊόν είναι καλύτερο. Και από ανθρωπιστικής και από οικονομικής πλευράς να δούμε τι θα γίνει. Άλλωστε αν υπάρξει απαγόρευση της μεταφοράς αυτό θα τονώσει στις τοπικές κοινότητες και την ε, Ήπεθρο και αν υπαγορευτούν μεταφορές θα γίνεται και κατανάλωση κοντά στο σημείο της παραγωγής. Αυτό όμως αν δεν θεωρείται ρεαλιστικό τότε θα πρέπει ρεαλιστικά να εφαρμόσουμε τον ε, κανονισμό. Οπότε παρακαλώ την Επιτροπή χρησιμοποιήστε όλες τις δυτικές αρχές, όλες τις αρχές που μπορείτε ούτω ώστε να υπάρχει ο έλεγχο παντού, να ελέγχονται τα φορτηγά, ούτω ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Ένα λεπτό η κυρία Χολ. Κύριε Επίτροπε, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε υπόψη της τις υγειονομικές συνέπειες από αυτή την νομοθεσία. Γιατί αυτές οι μεταφορές σε μεγάλη απόσταση φέρνουν αγωνία, στρες στα ζώα και μετά γίνονται πιο ευάλωτα όσον αφορά τις ασθένειες. Αυτό ισχύει και για τα ζώα. Υπάρχει ε, επιστημονική τεκμηρίωση ότι ε, τα ζώα αφοδεύουν πολύ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει γίνονται πιο τεταράλογα, ε, γίνονται πιο ευαίσθητα. Έχουμε 320 εκατομμύρια ζώα τα οποία μεταφέρονται προς το σφαγείο κάθε χρόνο και έχουμε βέβαια έτσι περισσότερες πιθανότητες για να πάθουμε σαλμονέλα. Μια που δεν εφαρμόζεται καλά αυτή η νομοθεσία ακόμα και με στάσεις, ιδίω τα άλογα ε, υφίστανται όλο αυτό το στρες μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει να λάβει υπόψη της αυτή την επιστημονική τεκμηρίωση να έχει κάποιο άλλο είδους ε, όρια μεταφοράς και έτσι να ωφεληθούν και τα ζώα αλλά και οι άνθρωποι. Ποντκάνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα αυτό της μεταφοράς είναι πολύ σημαντικό και άρα είναι πάρα πολύ θετικό το ότι τώρα εδώ καθόμαστε και τα ξανασυζητάμε. Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός όμως με τρόπο αποτελεσματικό. Επίσης, θεωρώ πολύ θετικό το ότι ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταφορά των αλόγων. Αυτό δεν το λέω βέβαια γιατί εκτρέφω εγώ ε, άλογα, αλλά σας το λέω και γιατί γνωρίζω ότι τα επιτασσόμενα από την νομοθεσία δεν εφαρμόζονται. Τα άλογα σας διαβεβαιώ μας νιώθουν, μας καταλαβαίνουν. Εμείς όμως δεν κάνουμε το ίδιο. Υπάρχει φόβος, υπάρχει εμπιστοσύνη, όλα αυτά τα συναισθήματα ε, που υπάρχουν και εγώ πολλές φορές έχω αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις ε, ακόμα και άρρωστα ζώα πολλές φορές ξέρετε οι ιδιοκτήτες τους δεν τα πηγαίνουν στον κτηνίατρο κάθονται και τα κοιτάνε οπότε φυσικά μετά και δυσπιστεί το άλογο προς τον άνθρωπο, ακόμα και προς τον κτηνίατρο. Θα πρέπει να συμπαρασταθεί ο ιδιοκτήτης προς το ζώο, θα πρέπει να πάει μαζί του στον γιατρό, τέλος πάντων δεν θα πρέπει να κάνουμε τα ζώα να υποφέρουν και θα πρέπει με όλα αυτά εμείς να τα καταλαβαίνουμε ως άνθρωποι. Έτσι γίνεται με τα ζώα, τα οποία μετά γίνονται επιθετικά όταν χάσουν την πιστοσύνη τους. Όμως, εάν φερθούν φιλικά οι ιδιοκτήτες, όλα αυτά αλλάζουν. Άρα θα πρέπει όλη η διαδρομή της εκτροφής του ζώου μέχρι το τέλος να είναι πιο ανθρώπινη. Τρία λεπτά τώρα. Ντελάνγκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε για άλλη μια φορά το θέμα της μεταφοράς των ζώων προσπαθώντας να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Η θείουσα νομοθεσία καθυστερεί στη σχέση με τις φιλοδοξίες που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως το είχαμε δει και στην έκθεση Τζελ Χαμάτ, που μιλούσε για τη διαφορά μεταξύ των ζώων που προορίζονται για σφαγή και άλλων τύπων ζώων. Έχουν ληφθεί ε, κάποια μέτρα για την καλύτερη ποιότητα των μεταφορών, για τη χρήση GPS κλπ. Αλλά δεν αρκούν αυτά τα μέτρα, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Και ο έλεγχος είναι η αχίλιος πτέρνα αυτών των συστημάτων. Δεν είναι εύκολο να γίνει ο έλεγχος σε ολόκληρη την Ευρώπη και βλέπουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικός και δεν είναι οργανωμένος κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν πολλά προβλήματα και κατά τη διέλευση των συνόρων και εγώ θα προτιμούσα να παρεμβαίνει πιο συχνά η ιατρική υπηρεσία Τώρα συζητάμε τις ε, εθνικές εκθέσεις ε, που πρέπει να υποβάλλονται και που θα πρέπει να αξιολογήσει η Επιτροπή. Είναι σαν να ανήπτει τα σχήρια τη η Επιτροπή. Θα έπρεπε όμω να φροντίσει η Επιτροπή να υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό έλεγχο, να υπάρχει επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί υπάρχουν δυνατότητε βελτίωση τη νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι χώροι ανάπαυσης με καλύτερο εξοπλισμό ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση και θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής σε μια τράπεζα δεδομένων. Δεν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις ε, στην ε, Αυστρία να, υπάρχει, να γίνεται κάποιος ε, έλεγχος όταν στην Αυστρία θα βλέπουν ότι φεύγουν φορτηγά προς τον νότο αν δεν εντοπίζονται τα ίδια φορτηγά μεταφοράς των ζώων στην Τσεχία θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία κάποιο σύστημα για να γίνεται σωστά τελικά η παραγωγή παρακολούθηση και να εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα τηρούν την νομοθεσία κατά τον ίδιο τρόπο. Και το θέμα των κτηνιάτρων ε, ε, είναι σημαντικό. Οι κτηνίατροι που επιβλέπουν τις μεταφορές δεν πρέπει απλώς να σφραγίζουν τα έντυπα, θα πρέπει να ασκούν έργο ελέγχου. Όταν μιλάμε για μεγάλες μεταφορές, ε, τα 500 χιλιόμετρα φαίνεται ότι χρειάζονται ε, δυόμιση ώρες ε, με, με βάση κάποια έγγραφα με Φεράρι τα μεταφέρουν τα άλογα αυτά. Ε, χρειάζεται κάποιος έλεγχος των στοιχείων που δηλώνονται. Πολλά είναι τα στοιχεία λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή. Έχει πολλή δουλειά μπροστά της και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις της πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Λίν, ένα λεπτό. Εγώ θα μιλήσω κυρίως ε, για τη μεταφορά των αλόγων, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν ε, στοιχεία που δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές διατάξεις ε, υπέρ της ευζοίας των ζώων και υπέρ των καλών συνθηκών μεταφοράς δεν τηρούνται και καταλήγουν σε μεγάλη τελεπορία των ζώων. Πολύ συχνά τα άλογα είναι σαν σαρδέλες μέσα στα οχήματα μεταφοράς και μπορεί να είναι μεταλλικά τα οχήματα μεταφορά του, πράγμα το οποίο αυξάνει υπερβολικά τη θερμοκρασία, οδηγεί σε θερμοπληξία και σε αφυδάτωση. Η Επιτροπή έχει φροντίσει ε, να εξετάσει το τι έχει γίνει με την τήρηση του κανονισμού 1 του 2005. Έχει οδηγήσει στο δικαστήριο κάποια κράτη-μέλη για τη μη τήρηση του κανονισμού από τότε που τέθηκε σε ισχύ το 2007 θα εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την παρακολούθηση των μεταφορών. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόσβαση της Επιτροπής σε κάποια δεδομένα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες. Θα ήθελα λοιπόν απάντηση από την Επιτροπή στις ερωτήσεις αυτές. Ο κύριος Ντόβερ, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά λαμβάνω το λόγο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που συζητούμε σήμερα και για αυτό και σας τονίζω ότι στη βορειοδυτική Αγγλία η μεταφορά των ζών των ζώων είναι τέτοια που δικαιώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας όσον αφορά τη μεταφορά και τη σφαγή τους. Πολλές φορές πρέπει να ακολουθεί μια τέτοια διαδικασία ε, μεταφοράς κλπ. μέχρι το τελικό προϊόν. 18 ε, ε, ε, χρόνια ως μέλος του Εθνικού μας Κοινοβουλίου. Έχω ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα επανειλημμένα, γιατί αυτό το πρόβλημα κρεμεί εδώ πολύ καιρό και δεν έχει υπάρξει τελευταία δεκαετία και 20 ετία κάποια εντυπωσιακή βελτίωση της κατάστασης. Γι' αυτό και χαίρομαι που ανεφεί το θέμα και το συζητούμε, διότι ξεκινήσαμε το 2007, Ιούνιο του 2006, έπρεπε 2008 έπρεπε να έχουμε την έκθεση, άρα έχουμε μείνει πίσω, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την δορυφορική παρακολούθηση της κατάστασης. Πάντως, ε, πολλές φορές Έχουμε ελέγχους που άλλωστε προβλέπονται και από τον κανονισμό. Για τον τρόπο μεταφοράς, για τα μέσα μεταφοράς, για τα κοντέινερ της καταθάλασσας μεταφοράς, τις στάσεις, το χώρο που θα πρέπει να προβλέπεται. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί τα δύο δορυφόρος, άρα χρειάζονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι ή αυστηρή. Όλα αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν και ελπίζω ότι τελικά ο Επίτροπος ε, θα μπορέσει όλα αυτά να τα λάβει υπόψη το νωρίτερο δυνατόν και έτσι να γίνει η εφαρμογή του κανονισμού. Και άλλωστε όσο νωρίτερα κινητοποιηθούμε τόσο καλύτερα γιατί είναι απαράδεκτο τα ζώα θα πρέπει στις τελευταίες μέρες της ζωής τους να έχουν τέτοιες συνθήκες μεταφοράς όπως θέλουν ε, τις κόντες ελεύθερης βοσκής και τα αυγά από αυτές τις κόντες οι καταναλωτές θέλουν αντίστοιχα και ανθρώπινη μεταχείριση προς τα ζώα. Ο κόσμος νοιάζεται για τα ζώα και θέλει να νοιάζομαστε και εμείς. Κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με την διατροφή μας. Ευχαριστούμε κύριε Ντόβερ, λέει ο Πρόεδρος. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Πόγεμο. Κύριε... Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κύριο Νίλ Πάρης για τη συζήτηση αυτή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το να διασφαλίσουμε σωστέ συνθήκε για τη μεταφορά των ζώων και θα πρέπει η Επιτροπή να φροντίσει να γίνονται οι σωστοί έλεγχοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια τη μεταφορά των ζώων. Υπάρχουν διατάξεις ε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχώς σοβαρές παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Υπάρχουν διατάξεις ε, που επαρκούν εφόσον βέβαια εφαρμόζονται και εφόσον γίνεται σωστά η παρακολούθησή τους και πρέπει να γίνεται σωστά η παρακολούθηση όλων των ε, διατάξεων αερισμού, θερμοκρασίας, ε, πυκνότητας των ζώων κατά τη μεταφορά, παρακολούθηση μέσω δορυφόρου. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται. Οι διατάξεις ε, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται σωστά και θα πρέπει πρώτα να φροντίσουμε την εφαρμογή πριν μιλήσουμε για την διατύπωση νέων κειμένων. Ευχαριστώ. ώρα Συνάδελφε, ευχαριστούμε. Και τώρα ήρθε η ώρα των ερωτήσεων το σύστημα Catch the και συνήθως ε, δίνουμε το λόγο μέχρι πέντε συνάδελφους. Το έχουν ζητήσει 7, αλλά έχουμε τα χρονικά περιθώρια, οπότε θα δώσουμε και στου 7 συνάδελφους το λόγο, πάντως να τηρήσουν τα χρονικά όρια. Πρώτη, πρώτη η κυρία Σίργουμπρο να έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μέσα σε μια κοινότητα θα πρέπει ε, ε, όλοι να τηρούν τις διατάξεις για να μπορεί να υπάρχει ομαλή συνεργασία και τήρηση των διατάξεων. Νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή ποιότητα του κρέατος για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυγχάνεται μέσω της, ε, των σωστών συνθήκων μεταφοράς των ζώων. Οι κακές συνθήκες μεταφοράς ε, ε, μειώνουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος και υπάρχουν ε, και επιστημονικά δεδομένα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για τις ε, διατάξεις μεταφοράς των ζώων. Θα πρέπει να τηρούν όλοι τις διατάξεις και οι μεταφορείς από τρίτες χώρες και θα πρέπει να επιβάλλονται οι κατάλληλες τιμωρίες αν δεν τηρούνται αυτές οι διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρμπετ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχουν σοβαρέ αμφιβολίες για το κατά πόσον η τρέχουσα νομοθεσία λειτουργεί ή όχι, κατά πόσον εφαρμόζεται ή όχι σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά ακόμα και σε περιπτώσει όπου μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία όταν, υπάρχουν, όταν έχουμε διεθνή μεταφορά των ζώων νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσον θα πρέπει να επανέλθουμε στην ιδέα ενός αυστηρού ορίου μεταφοράς 8 ερών χωρίς καμία εξαίρεση, εκτός βέβαια την, την μεταφορά διαθαλάσσης για τα νησιά. Αλλιώς να μην υπάρχει καμία άλλη εξαίρεση. Να σας πω ότι υπάρχει και ένα νέο website που, κάνει... που προωθεί αυτή την εκστρατεία, είναι www.8ώρες.eu το 8 ψηφία, όχι γράμματα. Τέλο πάντων, ίσω να, είσαστε, να ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την... Ε, να διαβάσετε το website αυτό και να δείτε τι λέμε. Ο κύριος Σούλτ. Κάπως έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε το ότι θα πρέπει να έχουμε ανθρώπινη, ανθρωπιστική συμπεριφορά για τη μεταφορά των ζώων που είναι πολύ σημαντική υπόθεση είναι πάρα πολύ σωστά τα όσα συζητήσαμε αλλά σας επισημαίνω ότι παρά το ότι έχουμε τη σωστή κατεύθυνση δεν θα πρέπει να έχουμε τεχνητούς φραγμούς ε, να επιβάλλουμε κάποια πράγματα που δεν είναι λογικά προς τους κοινοτρόφους και η Κομισιόν και όλοι μας ας λάβουμε υπόψη το ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική να μην είναι πάρα πολύ δίσκαμπτο το νομοθέτημα και βεβαίως η εξέβρεση λύσης είναι σημαντική υπόθεση όμως ας εξασφαλίσουμε όλοι ότι θα γίνει υπεύθυνη εφαρμογή του κανονισμού από όλα τα κράτη-μέλη. Ο Πρόεδρος. Κύριε Δημητρίου, έχετε το λόγο. Δημητρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η έρευνα για τα, πάνω στα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντική για την πρόοδο της βιολογίας και πρέπει να δούμε πώς ε, εκτρέφονται και πώς ζουν τα ζώα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει πάνω από 20 χρόνια που εφαρμόζεται και τα πράγματα εκεί είναι κατά προσέγγιση. Όμως έχουμε δει ότι πολλές χιλιάδες ζώα έχουν χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα η ευημερία των ζώων θα έπρεπε να αποτελεί μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία ζώων, η μεταφορά, οι, οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι θυσίες, οι σφαγές, όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται σε ευόμενη την διεθνή νομοθεσία έτσι ώστε να αποφεύγουμε την αγριότητα απέναντι ε, στα ζώα. Ο επόμενος Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα νέα κράτη-μέλη, και ιδιαίτερα θα μιλήσω για τη Ρουμανία, τη χώρα μου, χρειάζονται υποστήριξη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ε, την νομοθεσία και να πιέσουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων. Είναι ένα δύσκολο κείμενο για τις κτηνιατρικές αρχές της Ρουμανίας. Είναι δύσκολο το να ελέγξουν ε, τη μεταφορά των ζώων χωρίς ε, να ζητήσουν βοήθεια από την αστυνομία που είναι η μόνη αρχή υπεύθυνη ε, που θα, μπορούσε να σταματήσει ένα όχημα για να κάνει ελέγχους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η μεταφορά των ζώων από τα βουνά στις παιδιάδες που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Και επίσης ε, θα ε, ε, ήθελα να αναφέρω ότι η έλεγχοι και οι εκθέσεις που συζητάμε θα πρέπει να μας εγγυώνται το σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η κατάσταση του φορτηγού αλλά και οι ικανότητες του οδηγού και η συμπεριφορά του είναι οι προϋποθέσεις για την ευημερία των ζώων. Δεν οδηγάνε να κάνουν ράλι, να στρίβουν απότεμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, κακό για τα ζώα. Θα πρέπει να είναι σύγχρονο το φορτηγό και να οδηγείται με προσοχή. Αυτό ισχύει κυρίως και για τα άλογα που πάνε για σφαγή, γιατί πολλές φορές κάποια κράτη-μέλη ξέρουμε ότι επίτηδες δεν εφαρμόζουν την σχετική νομοθεσία. Έχετε την έκθεση από την Ιρλανδία που καταγγείλαμε επίτροπε τις χώρες που δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Αναλάβατε ενέργειες κατά αυτών των παραβατών. Παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ευχαριστούμε κύριε Αντώλιο Πρόεδρος και τώρα θα ολοκληρωθεί το Κατσιδιάδη με τον κύριο Σικιάστη που θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Όντω αποδείται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ευημερία των ζώων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να ισχύει από την ώρα που γεννιούνται μέχρι την ώρα που θα πάνε στο σφαγείο. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα πρέπει να ε, συνδέσουμε την ποιότητα του υλικού προϊόντος με την καλή μεταχείριση που έχει προηγηθεί πριν σφαγεί το ζώο. Γι' αυτό και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Πολλές φορές βέβαια χρειάζεται να ταξιδέψουν τα ζώα κάποια μεγάλη απόσταση για δηλαδή το οποίο απαιτεί χρόνο όμως θα πρέπει κατά όλο αυτό το διάστημα να τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις. Θα πρέπει να γίνει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας θα πρέπει να δούμε τι κάνει το κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να θυμόστε πάντα ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κάτι το δαπανηρό που μετακυλίεται ως εφαρμογή στον καταναλωτή. Κύριε Πάρης, θα σας δώσω λόγο μια που είστε πρόεδρος της ε, σχετικής επιτροπής, αλλά παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Πάρης, ναι, θα είμαι σύντομος πρόεδρε, ε, ε, γιατί θα ήθελα να το πω πριν συνοψίσει του κύριου Επιτρόπου, έχω εδώ πέρα κάποιε ερωτήσει που είχα υποβάλει, απάντησε την πρώτη για τα κράτη-μέλη που υπέβαλαν κάποιε εκθέσει και καταγγελίε. Έχετε κάνει κάποια προκριτική ανάλυση σχετικά με το πώ έχουν τα πράγματα. Πρόκειται εσεί να συντάξετε κάποια έκθεση σχετικά με το τι γίνεται με τον οργανισμό στο μέλλον. Αυτό χρειάζεται να ισχύσει η άριστη πρακτική. Έχουμε την Σλοβενία που παρακολουθεί τα φορτηγά. Μερικά κράτη έχουν καλέ επιδόσεις, μερικά άλλα είναι κακοί μαθητές. Θα κάτσετε να κάνετε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Και πότε, Επίτροπε, ο Πρόεδρος. Ωραία, ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Σπίτλα θα λάβει το λόγο. Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Το ρωμαϊκό δίκαιο στον ορισμό για τα ζώα ορίζει ότι ένα ζώο ε, είναι πράγμα. Θυμάμαι ένα στρατιωτικό κανόνα που για θέματα μεταφορών ε, έλεγε ότι σε ένα βαγόνι μπορεί να μεταφέρονται 8 άλογα ή 24 ε, άνδρες. Θεωρούμε σιγά σιγά με την πρόοδο του πολιτισμού ότι υπάρχει μεγαλύτερη σχέση μεταξύ ανθρώπου και ζώου παρά μεταξύ ζώου και πράγματος. Θεωρούμε ότι ένα ζώο δεν είναι πράγμα, είναι ένας οργανισμός που αναπνέει, που έχει δικαιώματα και αυτό το έχουμε εκφράσει στους αντίστοιχους κανονισμούς και διατάξεις. Υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αυτό τον τομέα και νομίζω ότι αποτελούν πρόοδο στο πλαίσιο της εξέλιξης του πολιτισμού μας. Βλέπουμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της συζήτηση που έγινε ότι οι διατάξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρούνται ευλαβικά και υπάρχει μεγάλος χώρος, μεγάλο πεδίο βελτίωσης. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι χρειάζεται βελτίωση και θα προσπαθήσει να βελτιώσει το σύστημα, να βελτιώσει τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις, την παρακολούθηση και παράλληλα Προετοιμάζουμε νέους κανονισμούς που θα λαμβάνουν υπόψη τις πλέον εξελιγμένες ε, επιστημονικές πληροφορίες από πολλούς τομείς. Διότι, όπως φάνηκε από τη συζήτηση αυτή, είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα όπου μπορούμε να κάνουμε ένα ή δύο πράγματα και θα έχουν ρυθμιστεί τα πάντα. Η συζήτηση έδειξε ότι η έννοια της προστασίας των ζώων, ιδίως των ζώων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία, δεν είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με την προστασία των καταναλωτών. Ορισμένα από τα μέτρα που συζητούνται θα πρέπει να ληφθούν ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν είχαν επιπτώσεις για τους καταναλωτές, απλώς και μόνο διότι είναι θέμα ηθικής και δεοντολογίας. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που έγιναν. Επειδή έγιναν πολλές ερωτήσεις, η Επιτροπή θα είναι πρόθυμη να απαντήσει περαιτέρω και μετά την σημερινή συζήτηση. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έγιναν. Όσον αφορά τις χώρες που έχουν στείλει την έκθεση, Ήδη το ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση. Θα επαναλάβω ότι ήταν η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο οι χώρες που δεν έχουν υποβάλει έκθεση αφού το θεωρήσατε τόσο σημαντικό. Δεν μίλησα για την Ιρλανδία λοιπόν. Η Ιρλανδία έχει εκπληρώσει το καθήκον της για την υποβολή έκθεσης. Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα της προσβασιμότητας σε πληροφορίες. Θεωρητικά είναι δυνατόν ε, οι εθνικές εκθέσεις να δημοσιεύονται. Ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ορίζουν και κάποια στοιχεία εμπιστευτικότητας, αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα καμία χώρα μέλος. Η Επιτροπή μπορεί να ρωτήσει λοιπόν τα κράτη-μέλη αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα της εμπιστευτικότητας και αν δεν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη θα μπορεί να δημοσιεύεται η έκθεση και να είναι προσβάσιμη ανοιχτά προς όλους. Πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα και σε περαιτέρω ζητήσεις. Οι αιτήσει εκθέσεις αναλύονται από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και συμπληρώνονται από τα στοιχεία τα οποία αποκτούμε από τους επιθεωρητές που έχουμε επιτόπου και αυτό δίνει δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονισμού και των περαιτέρω εξελίξεων του νομικού πλαισίου. Τώρα όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις και τις πιθανές προτάσεις που θα υποβληθούν για τροποποίηση. Είναι ένα θέμα το οποίο το επεξεργάζεται η Επιτροπή. Προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις Και επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχουν ε, διαδικασίες ε, παραβίασης ε, της νομοθεσίας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο τέτοιες διαδικασίες επί παραβάση. Έχουν υποβληθεί δύο ή τρεις καταγγελίες σε σχέση με την Ανδαλουσία στην Ισπανία και συνολικά έξι κράτη-μέλη ελέγχθηκαν το 2008. Αυτά είναι τα αριθμητικά στοιχεία που έχω σε σχέση με τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε που έδειξε ξεκάθαρα ότι οι θέσεις της Επιτροπής και οι απόψει των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αφίστανται και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλό μήνυμα για το μέλλον σε αυτό το πολύ ευαίσθητο τομέα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έτσι τώρα ολοκληρώνεται αυτό το θέμα μας και πάμε στο επόμενο σύμφωνα με τη μέρη διάταξη που αφορά μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει υποβάλει ο κύριος ε, Πάρης εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και η ερώτηση αυτή αφορά την μεσογειακή δίαιτα. Και τώρα.